διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών με ειδοποίησε ότι δεν έχει διατυπωθεί καμία αντίρρηση στη διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών στη σύσταση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής να μην διατυπωθεί αντίρρηση σχετικά με κατεξιοδότηση πράξη. Εάν δεν διατυπωθεί αντίρρηση στη σύσταση από μια πολιτική ομάδα ή από 40 τουλάχιστον βουλευτές εντός 24 ωρών, η σύσταση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Σε διαφορετική περίπτωση η σύσταση θα τεθεί σε ψηφοφορία. Η σύσταση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι